στο μέλλον, διότι είναι ένα μέσο το οποίο αποδεικνύει την ευρωπαϊκή ελληνική απέναντι στου εργαζόμενου που απολύονται. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Άρα τελειώνει εδώ πέρα η συζήτηση. Η ψηφοφορία είναι αύριο στις 12.30. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ακολουθεί τώρα η έκθεση του κυρίου Λέχνερ, διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων και τον λόγο έχει ο εισηγητή για 4 λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο σημαντικά είναι τα μητρώα των επιχειρήσεων, τα εμπορικά μητρώα ή όπως αλλιώς ε, λέγονται, φαίνεται από τις πάρα πολλές οδηγίες ε, που είχαν ξεκινήσει από το 1968 να ασχολούνται με αυτό το θέμα και βέβαια έχουν επιφέρει πάρα πολλές ε, βελτιώσεις. Το 2003 είχαμε μια ουσιαστική αλλαγή γιατί είχαμε πλέον υποχρέωση ηλεκτρονικών μητρών και αυτό οδήγησε στην καλύτερη διασυνοριακή πρόσβαση. Τώρα βεβαίως θα πρέπει να δούμε το ποιος είναι ο αρμόδιος για εθνική καταχώρηση σε εθνικό επίπεδο. Και βέβαια αυτό δεν θα αλλάξει. Όμως η πρόσβαση σε αυτό είναι σημαντική και πρέπει να βελτιωθεί και πρέπει να το τονίσουμε. Το πρόβλημα βεβαίω έχει δύο πτυχές. Η μία είναι η πρόσβαση για τους πολίτες, τους πολίτες που μπορεί να είναι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, ένα λογιστής, ένα μέλος ενός συνδικάτου, ε, ένα εργαζόμενος που θα πρέπει να βελτιωθεί στο, στη συνοριακή του πτυχή και βεβαίω το δεύτερο κομμάτι είναι η διαλειτουργικότητα, η συνεργασία μεταξύ των μητρώων που θα πρέπει να βελτιωθεί και αυτό αφορά κυρίως τις περιπτώσεις οποίες ε, μία επιχείρηση η οποία συναλλάσσεται σε μία χώρα με ένα υποκατάστημα και χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να έρθει σε επαφή με την έδρα με το κεντρικό κατάστημα μιας επιχείρησης, κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να γίνει πιο αυτόματα. Βεβαίως ε, όλοι χαιρετίζουν τις ε, άοκνες προσπάθειες της ε, Κομισιόν. Αυτό σημαίνει πως θα εξοικονομήσουμε κόστος και χρόνο και θα βελτιωθεί η εσωτερική αγορά. Να αναφέρω πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα, πως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες, γιατί τι σημαίνει αυτό. Έχουν νομική ισχύ η οποία όμως διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ αυτό οι χρήσεις για να μην έχουν την εντύπωση πως αυτό το οποίο ισχύει στη δική τους χώρα ισχύει και σε κάτι άλλο που διαβάζουν σε ένα άλλο μητρό. Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει όμως μια ομοιόμορφη μορφή για να υπάρξει μια ενιαία πύλη διαδικτυακή. Βεβαίως και εκεί πέρα μπορεί να λυθεί το γλωσσικό. Θα μπορούσαν να περιέχονται και όλες οι επίσημες γλώσσες. Υπάρχουν ήδη αρκετές πρωτοβουλίες γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο το EBR, το Bright, ε, τις πρωτοβουλίες δηλαδή για την διαλειτουργικότητα των μητρώων επιχειρήσεων, που όπως ε, συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι είναι πρωτοβουλίους θα πρέπει να εμφανιστούν βεβαίως ε, να εμβαθυνθούν έχουν όμως το μειονέκτημα ότι είναι πρώτον εθελοντικές, δεύτερον δεν συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις σε αυτό και τρίτον βεβαίω ότι βρίσκονται σε ένα στάδιο πειραματικό. Βεβαίω, εγώ και το Κοινοβούλιο δεν έχει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεν είναι και η δουλειά μας άλλωστε, οπότε εγώ θα ήθελα να προωθηθούν αυτές ε, οι πρωτοβουλίες. Αυτό είναι και ομόφωνη γνώμη των συναδέλφων και βεβαίως θα οδηγηθούμε σε επιτυχία μόνο εάν συμφωνήσουν όλες οι επιχειρήσεις να συμπεριληφθούν. Οπότε, εάν ε, λειτουργήσει κάτι τέτοιο θελοντικά δεν χρειάζεται καν και νομοθετική πρόταση. Οπότε καλό είναι να προωθήσουμε αυτή την υπόθεση όταν έχει οριμάσει βεβαίω και όταν θα συμμετέχουν και όλε οι επιχειρήσει και όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω και του συναδέλφου και τι επιτροπέ και υποθέτω νομίζω πω ε, θα εγκριθεί και ομόφωνα η έκθεσή μου πώ έγινε και στην Επιτροπή. Σα ευχαριστώ κύριε Λέχνερ. Έχουμε ξανά πέντε λεπτά συζήτηση με τη διαδικασία και έτσι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το λόγο έχει η κυρία Ρόιτοβα. Ε, Συνάδελφοι, τα μητρώα επιχειρήσεων δεν διασυνδέονται αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό αποτελεί αποτυχία της Κομισιόν, που είναι το συντονιστικό όργανο για χρόνια τώρα. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν εμπορικά μητρώα. 19 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και το δικό μου, ε, έχουν συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα μητρώων, αλλά η, σε ορισμένα κρατημέλη η ποιότητα αυτών των ε, μητρών δεν είναι η απαιτούμενη. Δεν καταγράφονται όλες οι επιχειρήσεις κλπ. Καλό λοιπόν την ε, Κομισιόν να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το φαινόμενο. Και τα υπόλοιπα οκτώ πρέπει επίσης να υποστηρίξουν οικονομικά αυτό το project και να συμμετάσχουν. Είναι πολύ σημαντική η ε, πρόσβαση, διασυνορική πρόσβαση. Όχι, η κυρία Ρέγνερ τελικά έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λέχνερ για την καλή συνεργασία πρακτικά βρέθηκαν όλες οι συμβαστικές ε, λύσεις. Ε, εν ολίγης τώρα τα σημαντικότερα σημεία είναι βεβαίως ε, η συνδυσμευτική συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε αυτό. Δεύτερον, να υπάρχει μία δημόσια πρόσβαση από ένα επίσημο πόρταλ. Τρίτον, βεβαίω η προστασία των καταναλωτών που είναι ιδιαίτερα σημαντική, δηλαδή να είναι αξιόπιστες και επίκαιρες οι πληροφορίες και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ε, καταναλωτές γιατί βεβαίως εδώ πέρα υπάρχουν ε, και οι ένομες συνέπειες για τις οποίες θα πρέπει να είναι πληροφορημένες και βέβαια το σύστημα θα πρέπει να είναι πρακτικό και φιλικό προς τον ε, χρήστη. Αυτό πρέπει να είναι αποστολή της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ και τώρα έχει τον λόγο η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. την Ευρώπη των 27 ε, κρατών μελών, το 80% των, ε, μικρομεσαίων, των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η διασύνδεση των μικρών των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Από το... Ε, κοιτάξτε, ε, θα γίνεται ηλεκτρονική αποθήκευση και θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση όλοι σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά όμω, πρέπει να δούμε το θέμα των προτύπων. Ε, η γλώσσα, η μηχανή αναζήτηση, οι συνθήκε αναζήτηση είναι διαφορετικοί. Ε, γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε σχέδια όπως για παράδειγμα ε, η διαλειτουργικότητα των μητρών επιχειρήσεων, των εμπορικών μητρών, να η συμμετοχή σε όλα αυτά τα συστήματα ενημέρωσης ε, που αφορούν την εσωτερική αγορά. Διότι αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων ε, πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ε, και αυτή η εξοικονόμηση θα μπορεί να είναι ακόμα η μεγαλύτερη αν η πρωτοβουλια η e-invoices, δηλαδή η ηλεκτρονικά τιμολόγια, γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ κυρία Μπένοβα. Yeah. Vielen Dank. pani Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε πως ε, οι δυνατότητες ε, του εμπορίου απαιτούν την εναρμόνιση των δεδομένων ε, στα μητρώα αυτά. Είναι πλέον απολύτως απαραίτητο. Εάν τα καταφέρουμε να συνδέσουμε τα μητρώα των επιχειρήσεων, θα βοηθήσουμε και θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή και στις επιχειρήσεις αλλά και θα ενισχύσουμε την θέση τους γιατί βεβαίως θα υπάρχει και ασφάλεια δικαίου και, και διαφάνεια και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη για να είναι πολύ μεγαλύτερη η διαφάνεια και να έχουμε καλύτερη χρήση των δεδομένων για να δούμε παραδείγματο χάρη τι γίνεται όταν αλλάζει η έδρα μιας επιχείρησης όταν ιδρύονται ε, υποκαταστήματα σε άλλες χώρες όταν έχουμε συγχωνεύσεις λοιπά. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κιλ Νίλσεν. Ζητήσατε τον λόγο? Όχι. Ωραία. Εντάξει, γλιτώνουμε και λίγο χρόνο. Αμέσως λοιπόν ο κύριος Επίτροπος έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων είναι χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση τη διαφάνεια των οικονομικών εταίρων για την αποκατάσταση εμπιστοσύνη και την προώθηση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά. Συγχαίρω τον κύριο Λέχνερ και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την έκθεση αυτή. Συμφωνούμε ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό με την έκθεση αυτή και η Επιτροπή ε, το πολύ μέχρι τι αρχέ του 2011 θα υποβάλει νομοθετικέ ε, προτάσεις που σίγουρα θα λάβουν υπόψη συμπεράσματά σα. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε την ανάγκη ύπαρξη διαφάνειας στην χρηματοπιστωτική αγορά αλλά και πέραν τη αγορά, αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε επίσημα και αξιόπιστα στοιχεία ως και επικαιροποιημένα όσον αφορά τις εταιρείε. Και εδώ η διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων θα δίνει πληροφορίε για τι επιχειρήσει και βεβαίω οι πληροφορίε αυτέ ε, θα είναι προβάσιμε στο πλατή κοινό. Ε, γιατί συχνά ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τεχνικού λόγου ή γλωσσική φύσεω να ε, τι πληροφορίε ε, που έχουν οι πολίτε ενό κράτου μέλου το οποίο είναι εγκαταστημένη μια επιχείρηση να τι έχουν και οι υπόλοιποι. Η διασύνδεση λοιπόν θα αποτελέσει ένα πλέον εργαλείο υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των εργαζομένων. Τώρα, ε, να σα εκφράσω ορισμένε σκέψει όσον αφορά ορισμένε πτυχέ τη έκθεση του κυρίου Λέχνερ. Σημειώνω τι ανησυχίε σα σχετικά με το συμπληρωματικό διοικητικό άχθο που θα μπορούσε να είναι απόρρια τη διασύνδεση των μητρών αυτών. Μπορώ όμω να σα διαβεβαιώσω ότι ε, επουδενή λόγο δεν, πρόθεσή μα δεν είναι να επιβάλλουμε άμεσα ή έμεσα ε, επιπλέον κόστη στις επιχειρήσεις. Συμφωνώ με το ότι ε, η συμμετοχή όλων των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η ε, συμμετοχή στο μηχανισμό συνεργασίας. Και βεβαίως αυτός ο μηχανισμός θα έχει νόημα μόνο εάν τον υποστηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τη συνεργασία στα πλαίσια τη τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών, σε, ε, σχετικά με τις θηγατρικέ και τα υποκαταστήματα στο εξωτερικό, έχει την πρόθεση η Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση ε, για ένα τέτοιο μηχανισμό. Και εκεί θα πρέπει να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη. Πρόκειται ε, για κάτι το οποίο λείπει στα πλαίσια της εσωτερική αγοράς. Επίση, υποστηρίζεται την υλοποίηση ενό ενιαίου σημείου πρόσβαση τη πληροφορία. Συμφωνούμε με το στόχο ε, τη προσβασιμότητα στα δεδομένα, ε, τα οποία υπάρχουν στα εθνικά μητρώα. Οι καταναλωτέ, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά και οι εθνικέ διοικήσει των άλλων κρατών μελών θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβαση στι υπηρεσίε αυτέ χωρί κανένα εμπόδιο. Κάτω από την ίδια αυτή οπτική γωνία τη ε, προσβασιμότητα, θέλουμε να προσφέρουμε πληροφορίε σε όλε τι επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ, ε, αυτό αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για την επίτευξη του στόχου τη προσέγγιση ε, τη ιστορική αγορά στου πολίτε. Εξάλλου, οι χρήστε των μητρών θα πρέπει να είναι απόλυτα ενήμεροι για τι συνέπειε των εθνικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στα μητρώα, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ανάλογα με το κράτο μέλο. Όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων, είναι σαφέ ότι οι πληροφορίε που παρέχονται στα πλαίσια τη διασύνδεση θα πρέπει να είναι αξιόπιστε, επικυρωποιημένε και προσπελάσιμε. Πρόκειται για κάτι σημαντικό. Ε, ε τονίζετε εσεί με αποφασιστικότητα το μήνυμα αυτό και εμεί με την ίδια αποφασιστικότητα βλέπουμε το θέμα αυτό. Σα ε, διαβεβαιώνω ότι κάθε προσπάθειά μα ε, θα σέβεται απόλυτα τα προσωπική φύσεω ή εμπορική φύσεω στοιχεία. Κυρίε και κύριοι, η έκθεση Λέχνερ δείχνει τη μεγάλη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ την κατεύθυνση τη υλοποίηση μεγαλύτερη διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων προ όφελο των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Το σχέδιο αυτό θα ενισχύσει στην εσωτερική αγορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή τη για το γεγονό αυτό. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την έγκριση τη έκθεση στην Ολομέλεια. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τελείωσε λοιπόν η συζήτηση. Η ψηφοφορία αύριο στις 12.30. Τώρα περνάμε στην έκθεση ΒΙΦΚΑ για την διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ουσιαστικέ και εμπορικέ υποθέσει.